colleagues, may I have your attention, please? Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε την καλοσύνη. Καθίστε. For members of the Econ Committee, um, my name is Claude Moraes. I'm chair of the Libe Committee. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τέβα, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών. Μωράες, και παρακαλώ πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε να ελέγξουμε αν έχουμε τις κάρτες για την ψηφοφορία. Ας κάνουμε αυτό τον έλεγχο πριν ξεκινήσουμε. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, λέει ο συμπρόεδρος κύριος Σιμών, ε, πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο Τοποθετήστε λοιπόν παρακαλώ τις κάρτες σας στο μηχάνημα και ψηφίστε όπως θέλετε, υπέρ κατά αποχή, για να βεβαιωθούμε μόνο ότι δουλεύουν σωστά. Πέρας της υποφορίες παρακαλώ. 59 υπέρ, 3 κατά, 16 εποχές, 78 ψηφίσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Το άρθρο 73.5 που σχετίζεται με τις δύο προτάσεις που έχουμε ονοποιών μας λέει το εξής και διαβάζω. Άρθρο 73.5 του κανονισμού. Εάν υπάρχει ανάγκη για συμβιβασμό πάνω σε ένα κείμενο ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια επιτροπή και υποβάλλεται το συμπεφωνημένο συμβαστικό κείμενο ε, εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για έγκριση. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε τα δύο κείμενα. Ξεκινούμε με την ε, ψηφοφορία στις εκθέσεις Κάρνης και Σαρσεντίνη. Και αν δεν θέλουν οι συγγητές να μιλήσουν πριν την ψηφοφορία, αρχίζουμε αμέσως. Μήπως θέλει όμως η κυρία Σαρσεντίνη. Παρακαλώ. Κλοντ. Πάλι σήμερα το πρωί στη Λίμπαξ, στη Λίμπαξ το σημαντικότερο. Να ευχαριστήσω δηλαδή τους σκιώδεις ηγητές και τον συνεισηγητή, τον κύριο Κάνης και το προσωπικό των δύο επιτροπών που μας βοήθησε σε αυτή τη ε, διαδικασία. Χρειάστηκαν δύο χρόνια από όταν ήρθε στο Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα για να φέρουμε την πρόταση αυτή και να την περάσουμε τελικά και νομίζω πως το Κοινοβούλιο με το Δημόσιο Αυτό Αρχείο βελτίωσε την πρόταση και κατάφερε να εργαστούμε όχι μόνο κατά του ξεπλήματος χρήματος ε, και της ε, τρομοκρατίας αλλά και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάρενς, ε, έχετε να πείτε κάτι, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά ευχαριστώ. Ξέρω πως μας αρέσει να ακούμε ο ένας ε, τον, τις ομιλίες του άλλου, ήταν ε, πραγματικά μια συναρπαστική διαδρομή, η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών μας ήταν δύσκολη και έγινε κάπως λιγότερο δύσκολη όσο περνούσε ο χρόνος. Αν είχαμε άλλους έξι μήνες ε, θα είχαμε συγχρονιστεί έντελος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, χρειάστηκαν πέντε τριμερείς διάλογοι. Το πρόβλημα δεν ήταν βεβαίω στο κοινοβούλιο ήμασταν ενωμένοι, η δυσκολία ήταν το συμβούλιο. Και εδώ πέρα οφείλω να ευχαριστήσω την ε, Ιταλική Προεδρία για τις ε, τεράστιες ε, προσπάθειες που έγιναν να βρεθεί ένας συμβιβασμός για μια ισορροπία σε σχέση με αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε ως νομοθετικό σώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εξ ονόματος των δύο επιτροπών σας ευχαριστώ ε, για την σκληρή δουλειά που κάνατε. Επί τη διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο την διαδικασία της ψηφοφορίας. Χρειάζεται πλειοψηφία σε κάθε επιτροπή χωριστά ή μια πλειοψηφία των ε, επιτροπών. Κοινή, κοινή πλειοψηφία λέει ο Πρόεδρος πλειοψηφία του συνόλου. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Προφανώς έχετε τις κάρτες σας μαζί. «45» είναι η πλειοψηφία. Ονομαστική ψηφοφορία. 45 ε, η πλειοψηφία επί του συνόλου. Νομίζω ότι θα περάσει, νομίζω ότι θα περάσει. Να δούμε. Ίσως τσίμα τσίμα. Έτσι είναι το χιούμορ της Επιτροπής μας. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Για το θέμα Κάρινς και Σαρτζεντίνη, για το ξέβλημα χρήματος. 87 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Γίνεται λοιπόν δεκτό. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία. Σάιμον και Κέρκοπ είναι οι εισηγητές. Θέλετε τον λόγο, οι εισηγητές. Ευχαριστώ τον κανονισμό για τη μεταφορά κονδυλίων. Τα ζητήματα είναι λιγότερο επίμαχα όσον αφορά βεβαίως σε σχέση με την ε, οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες που συλλέγονται όσον αφορά αυτούς που πληρώνουν και αυτούς που λαμβάνουν. Ε, είχαμε δύσκολες τεχνικές συζητήσεις, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Και νομίζω απεδόθη η ιδέουσα σημασία. Ο κ. κέρκοπ Συμφωνώ και εγώ με τις παρατηρήσεις και να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία. ευχαριστώ κύριε Κέρκο, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Λοιπόν, να ξεκινήσει ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 83 υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Ε, ε, γίνεται δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα πάει στην Ολομέλεια λοιπόν το κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Τελειώσαμε με αυτό.